Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι διαθέσιμα. Έχετε κάποιο σχόλιο. Όχι, θεωρούνται λοιπόν από